πρόσωπο να παίξει σημαντικό ρόλο στη διάσκεψη της Μαδρίτης και να διατηρήσει υψηλό επίπεδο της ε, Πρωτοβουλίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις σχέσεις με Ελληνική Μερική. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Σαλαφράγκα. Η συζήτηση ολοκληρώθηκε. Η εξοφορία θα διεξαχθεί στην πρώτη σύνοδο του Μαΐου. Σε ό,τι αφορά την μίληση διάταξη της ε, αυριανής συνεδριάσεως Τετάρτης, σας προτείνω σε συμφωνία με τις πολιτικές ομάδες να μεταθέσουμε σε μια προσεχή συνεδρίαση την έκθεση Κοτσολίνο για την προστασία των δημοσιονομικών ε, συμφέροντων ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την καταπολέμηση της απάτης. Υπάρχουν παρατηρήσεις περί αυτού. Όχι. Η τροποποίηση της σημερινής διάταξης ως εκ τούτου έγινε δεκτή. Σύμφωνα με μέσα διάταξη, τώρα περνάμε στην δήλωση τη ε, ύπαρξη εκπροσώπου τη Ευρωπαϊκή Ένωση για θέματα εξωτερική πολιτικής και Πολιτική Ασφάλεια, αντιπροέδρου τη Επιτροπή, κυρία Άστον, σχετικά με το Κυργιστάν.